μερίδιο των εσόδων από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Και επίσης ε, πρέπει να έχουμε ε, ε, και άλλες πηγές διασυνοριακών συναλλαγών κλπ. Ελπίζω να μην προδώσει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πολίτες. Η ανάπτυξη της υπαίθρου οι παραμεθόριες περιοχές. Όλες αυτές οι περιοχές θα πρέπει να έχουν ευκαιρία για ανάπτυξη. Και αυτό είναι, ευκαιρία, είναι υποχρέωση του Συμβουλίου. Αν δεν ανταποκριθεί θα απορρίψουμε την πρότασή του. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Η κυρία Γκουάρια Θαβάλ Ρουιάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και δύο χρόνια μιλάμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και τώρα που έφτασε η ώρα της αλήθειας δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Γιατί ο κύριος Μισελ δεν ήθελε να, θε φτάστηκαν, μέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί και όλα τα νέα που μα φτάνουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι θετικά. Αν αυτές οι συγκεντρώσεις αφορούν τα δεκαδικά που θα δώσουμε εδώ και εκεί και τι μπορεί να εξοικονομήσει το Συμβούλιο, σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο θα απορρίψει αυτή την πρόταση το, στις 20 Φεβρουαρίου πρέπει να συζητήσετε τι πολιτικές θέλουμε να προωθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα τις χρηματοδοτήσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να κάνουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί τα αποτελέσματα είναι καλύτερα αν γίνουν σε επίπεδο Ευρώπης αυτές τις πολιτικές παρά σε εθνικό επίπεδο. Γιατί είναι πιο αποτελεσματική η Ευρώπη. Γιατί μειώνονται οι ανισότητες, υπάρχουν υπάρχει περισσότερη αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη είναι η μόνη λύση σε όλες τις περιπτώσεις, αν κάνουμε ε, ευρωπαϊκές λύσεις, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Όλοι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί οι συζητήσεις στο Συμβούλιο γίνονται ε, με βάση λάθος αφετηρία. Αυτό που με απασχολεί είναι η πολιτική συζήτηση. Πώς θα καταλήξουν όλες αυτές οι συμφωνίες και όλες αυτές οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Το Green Deal, Πώς θα το χρηματοδοτήσετε. Αν κάποιοι από σας πιστεύετε ότι η μετάβαση προς μια ε, οικονομία ουδέτερη σε διοξίδιο το άνθρακα, πώς θα γίνει, πώς θα, αν δεν στηρίξετε τους γεωργούς, αν δεν στηρίξετε τις ε, ε, επιχειρήσεις, τις περιφέρειες, τους εργαζόμενους, υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω μόνο το εξή. Εάν δεν έχουμε ένα λογικό προπολογισμό, η εναλλακτική είναι οικονομική αδυναμία, πολιτική αδυναμία και κατακαιρματισμός του ευρωπαϊκού εγχειρήματος διάλυση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό, κύριο Κέρνερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι περισσότεροι από εμά μιλάμε για μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Εγώ λέω ότι πρέπει να πούμε καλύτερο προϋπολογισμό με βάση προτεραιότητες δαπάνες με προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη μια, ε, ο εργαζόμενος σε μια επιχείρηση ανησυχεί για τη θέση εργασίας του, ε, θέλει ε, νέες δεξιότητες ε, ψηφιακές που θα τον βοηθήσουν να διατηρήσει την εργασία του. Ε, επίσης, οι πολίτες ανησυχούν για την τρομοκρατία. Ε, θέλουν χρηματοδότηση Frontex, Europol για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης, οι φοιτητέ, οι εκπαιδευόμενοι στην Ευρώπη θέλουν το Εράσμους γιατί μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη, να γίνουν ε, μέλος, με, μέρος της. Πρέπει λοιπόν οι δαπάνες να είναι ε, σωστές Καμιά φορά τα κράτη-μέλη πρέπει να σκεφτούν πού θα γίνουν και εξοικονομήσεις. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και να το συζητήσουμε. Είναι ξεκάθαρο ακόμη ότι δεν πρέπει να γίνουν εκπτώσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Πολλές φορές ε, χρησιμοποιούνται ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ καταπατούνται οι ευρωπαϊκές αξίες. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας στιβαρός μηχανισμός ελέγχου που, δεν θα, που θα ανθίσταται στα πολιτικά παιχνιδάκια. Θα πρέπει το κράτος δικαίου να τηρείται, αλλιώ δεν θα δίδονται τα χρήματα. Αυτό άλλωστε περιμένουν και οι φορολογούμενοι. Τη σωστή χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ο κύριο Βιλίμσκι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πολλοί είναι οι φανατικοί οι οποίοι ε, ζητούν περισσότερα δύση για την Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι σωστή αντίδραση αυτή. Ε, η Βρετανία, μια μεγάλη χώρα, μας εγκατέλειψε και τώρα ζητάμε περισσότερα χρήματα, ενώ η Ένωση είναι μικρότερη, άρα χρειάζεται και λιγότερα κονδύλια. Και επίσης δεν απαντήσατε στο ερώτημα αν θα μετά φερθούν περισσότερες αρμοδιότητες στις Βρυξέλλες ή αν θα πάνε προς τα κράτη-μέλη. Αυτό το ερώτημα από το 2016 δεν είχε απάντηθη. Μετά το δημοψήφισμα για τον Brexit είχαν ε, υποβληθεί από την Κομισιόν πολλά σενάρια χωρίς να δοθεί απάντηση. Τώρα το 2020, στην ε, ε, ενδεκάτη μετά από μία τετραετία, αρχίζει μια διάσκεψη για το μέλλον, που δεν αρχίζει στο τέλος, στην αρχή του χρόνου, αλλά στη μέση του έτους και θα πάει και μέχρι το 2021. Το ζήτημα ε, αυτό της απέτηση για περισσότερα κονδύλια είναι περιττό αν δεν ε, προδιαγράψουμε τη μελλοντική κατεύθυνση της Ένωσης. Στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, υπάρχουν σχετικά, σχετικές προβλέψεις. λιγότεροι επίτροποι, για παράδειγμα, λιγότερες οδηγίες, λιγότερη, λιγότερη γραφειοκρατία. Εγώ ε, ως πολίτης ε, μιας χώρας που είναι καθαρός ε, χρηματοδότης δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω ούτε ένα σεν παραπάνω για αυτόν τον προϋπολογισμό. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Κορμόν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τον προπολογισμό είναι μια συζήτηση που αφορά το μέλλον μας. Ε, βεβαίως είναι μια τεχνική συζήτηση που καμιά φορά ε, αποθεί τον πολίτη. Γι' αυτό θα είμαι κάπως απλός για να μην αγνοήσουμε το διακύβευμα. Ο προπολογισμό για τα, τα πέντε προσοχή χρόνια θα επιτρέψει στην Ευρώπη ή όχι να ανταποκριθεί στην κλιματική πρόκληση και τις κοινωνικές επιταγές. Άρα θα πρέπει να είναι ένας μαχητικός προπολογισμό. Ένας σφαιρικός προπολογισμό ο οποίος ε, θα ευξήσει σε 1,3% ε, του ΑΕΠ προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να πραγματοποιήσει την οικολογική μετάβαση. Ένας μαχητικός προπολογισμό όπου τουλάχιστον 50% θα διατίθενται στην προστασία του περιβάλλοντος. Ένας μαχητικός προπολογισμό προκειμένου να έχουμε τα δημοσιονομικά εργαλεία υπέρ της δικαιοσύνης και της οικολογικής ε, μετάβασης φορολογώντας τις εκπομπές ε, του άνθρακα κυροζίνη κλπ. Αυτοί οι φόροι θα μπορέσουν να καταλήξουν σε, στην αύξηση δύο πόρων. Για δύο ευρώ αυτών των φόρων, ένα ευρώ θα πάει στα εθνικά ταμεία και ένα ευρώ θα πάει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έτσι θα σηματοδοτήσουμε τη βούληση να εξάλθουμε από αυτό το διέξοδο. Θα πρέπει να κινηθούμε προς, αυτή, προς αυτό το δρόμο. Είναι αναγκαστικό. Ε, κύριος ε, Ζιλ, ε, Κυρία Πρόεδρε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, δεν θέλουν πλέον να πληρώνουν το 1% του ΑΕΠ, αλλά θέλουν παρόλα αυτά να αποφελθούν από την Ευρώπη. Αυτό δεν λειτουργεί. Στην, ε, ε, στις ΗΠΑ ο προπολογισμό καταρτίζεται εντελώ διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης δυστυχώς υπάρχουν αντιπαραθέσεις από παλιότερες χώρες της συνοχής ή ζητήματα γεωργικής πολιτικής. Εάν όμως χρηματοδοτείται η στρατιωτική πολιτική, ε, καλύτερα να χρηματοδοτείται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ο, η φιλόδοξη χρηματοδότηση του προπολογισμού για την ε, συνοχή Εάν υπάρξει εδώ μια περιστολή της τάξης του 25%, οι κάτοικοι αυτών των ε, χωρών θα βρεθούν σε πολύ δεινή θέση. Πολύ χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκούσμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ε, δεν, η Κομισιόν και το Συμβούλιο ήρθαν σήμερα εδώ για να ε, ανακοινώσουν περικοπές στην πολιτική συνοχή και στην ΚΑΠ. Παραπλανούν τους πολίτες για την Πράσινη Συμφωνία ε, και προϊονίζονται όλα αυτά θεσμική κρίση. Οι προτάσεις αφορούν περικοπές σε σημαντικές ε, πολιτικές. Εμείς ε, θέλουμε να προχωρήσουμε τις ε, νέες πολιτικές, αλλά βλέπουμε πάρα πολλά έργα που διαιωνίζουν την χρήση ορυκτών καυσίμων ή περιορίζουν άλλες πολιτικές δημοσιονομικά δεν υπάρχει δυνατότητα να επενδύσουμε για να καλύψουμε κοινωνικές και οικολογικές ανάγκες. Δεν θέλουν να επενδύσουν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Μουρισάν, ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχήν να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι απουσιάζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τις προτεραιότητες της Κομισιόν από πέρσι, ιδιαίτερα αυτές που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσουν την αλληλεγγύη, ε, να χτίσουν το κοινωνικό πυλώνα. Ε, θα ήταν ε, πολύ δυσάρεστο να καθυστερήσει η έγκριση του προπολογισμού ή να μην προβλεφθούν επαρκή κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν του στόχους. Η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί σωστή ισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων προτεραιοτήτων και νέων στόχων. Οι νέοι στόχοι, ιδιαίτερα αυτοί που αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης θα ε, ολοκληρωθούν αν οι παλιοί στόχοι της συνοχής ολοκληρωθούν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να, να, να λειτουργήσει με οικονομικές και δομικές διαφωνίες. Θα πρέπει να καταργηθούν ή να μειωθούν. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με θαραλέα προς το μέλλον αν υπάρχουν διαφορές μισθών μεταξύ κρατών μελών και άλλες διαφορές. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς συνοχής και το, ε, να καταπολεμήσουμε την διαφθορά. Ευχαριστώ κύριε Μουρασάν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η προετοιμασία του επόμενου προϋπολογισμού ε, είναι ένα σημαντικό θέμα. Ο κύριο Σάρλ Μισελ έπρεπε να είναι εδώ. Αν δεν είχε τίποτα να μα πει, ας ερχόταν να καθίσει και να μα ακούσει. Γιατί η τελευταία ε, λέξη θα ελεγχθεί από το Κοινοβούλιο. Θα εγκρίνουμε τον προπολογισμό μόνο αν οι προτεραιότητέ μα είναι μέσα. Ποιε είναι οι προτεραιότητε, Πρώτον, συνοχή ε, ε, ΚΑΠ. Συνεχίζουν να είναι σημαντικά όλα αυτά στην Ευρώπη. Νέε προτεραιότητε τη Ένωση στο φω των πολιτικών μα φιλοδοξιών. Η Κομισιόν ζήτησε υποστήριξη τις προτεραιότητες που προσανατολίζονται στο μέλλον. Προϋπολογισμός για την έρευνα. Ε, μειώνεται κατά 500 εκατομμύρια ε, ευρώ. Η έρευνα είναι σημαντική λέμε και το είναι αυξάνουμε κατά 700 ε, εκατομμύρια. Θα πρέπει να επενδύσουμε εκεί που έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει να μειωθεί το οράσμος. Δεν θα πρέπει δηλαδή να παίξουμε τη μία πολιτική σε βάρος μιας άλλης. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι η μόνη θέση που μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε σωστά αυτά που συμφωνήσαμε. Είναι η, προ... η μόνη θέση που επιτρέπει στην Επιτροπή Φόντερ Λάιν να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στι διαπραγματεύσεις. Ε, ε, αλλιώς ε, θα απορρίψουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Και πρέπει να πω σαφώς ότι αν πρόκειται να επιλέξουμε μεταξύ δίμηνης καθυστέρησης και κακού προϋπολογισμού, θα προτιμήσουμε να ε, καθυστερήσουμε για δύο μήνες και εμείς ε, αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε από τον Νοέμβριο του 2018, να σταματήσει να σέρνει τα πόδια το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κυρία Γκουαλμίνη. Να μισή λεπτό. Είναι ώρα να, ε, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. αυτό το πολιετές είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων την επόμενη επταετία. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όλοι οι πολίτες περιμένουν ε, βελτίωση των πολιτικών. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο, στο 1,3 για να χρηματοδοτήσουμε την πράσινη συμφωνία δεν πρέπει κανείς να τολμήσει να αφαιρέσει από τα παιδιά τα βασικά τους δικαιώματα, ε, τροφή, υγεία, παιδεία, ε, τα παραδοσιακά προγράμματα ε, πρέπει επίσης να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχτούμε μείωση της πολιτικής συνοχής, της ΚΑΠ, του Εράσμους. Από την πλευρά των εσόδων ας σκεφτούμε και τον ψηφιακό φόρο και ε, την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογία εταιριών, ε, ένα μερίδιο και από εκεί. Πιστεύουμε σε περισσότερη Ευρώπη, όχι σε λιγότερη Ευρώπη. Πιστεύουμε στις ε, δημόσιε επενδύσει, όχι στην υποβάθμισή του, στη μείωσή του. Πιστεύουμε σε μια καλή κοινωνία που είναι η κοινωνία των πολλών και όχι των λίγων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν υποχρεούται να ακούσει τη φωνή μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Αρμόν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να προσεγγίσω τρία θέματα που αφορούν το Ταμείο Συνεχής. Καταρχήν τον όγκο αυτών των ε, ταμείων. Αν ε, η, η Ρουμανία απορροφήσει 60 ευρώ, οι επενδύσεις δεν θα είναι σημαντικές. Δεύτερον, ε, τα ποστά της προχρηματοδότησης. Αν έχουμε μία αύξηση ε, του ποσοστού προχρηματοδότησης, ορισμένες χώρες θα πρέπει να παρετηθούν από το Ταμείο Συνοχής. Τρίτον, ε, η διάρκεια εντός της οποίας θα πρέπει να ε, ε, απαιτηθούν οι πληρωμές σε ένα πλαίσιο που θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε σχέση με τον παρόντα προπολογισμό, αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τα ποστά απορρόφησης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μπορκία, για ένα λεπτό. Παίζουμε κάθε τόσο, είμαστε παρόντες σε αυτό το παιχνίδι. Πώς θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Αλλά σήμερα χρειάζεται ρεαλισμός. Δεν είδα ρεαλισμό σήμερα το πρωί. Είδα ευχές για βελτιώσεις. Μίλησαν διάφοροι για προπολογισμό που θα πρέπει να μειώσει τη, τη ρήπανση, τις ανισότητες, την ανεργία ένα μακρό ευχολόγιο. Αλλά μιλάμε για διαχείριση των δημόσιων πόρων. Πρέπει όποιος ε, διαχειρίζεται τους δημόσιους πόρους να σκέφτεται τις ε, σπατάλες και τις δαπάνε. Πρέπει να προωθήσουμε τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές, την έρευνα, την κοινοτομία, την γεωργική πολιτική. Αλλά όταν πρόκειται για να περικόψουμε πόρους ας πούμε, για να τις δώσουμε σε εθνικές ε, πρεσβείες ε, για να διαχειρίζονται διάφορα πράγματα ή για να τα δώσουμε για την Τουρκία, ε, τότε νομίζω ότι το πράγμα και η κουβέντα γίνεται περίεργη. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. ορισμένοι υπερασπίζονται στο Συμβούλιο το Ταμείο Συνοχής, άλλοι το Ταμείο Γεωργίας. Αλλά πού είναι η θεμελιώδη συζήτηση περί εξυγχρονισμού, η συζήτηση ότι πραγματικά προετοιμάζουμε την οικονομία μας για ένα Green Deal, η συζήτηση για τα, τους θεμελιώδες κανόνες του κράτους δικαίου. Πού βρίσκεται η συζήτηση. Και θα ήθελα να πω ότι αυτές ε, οι χώρες που λένε μεγαλοσχήμωνα λόγια, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, οι κάτω χώρες, ε, η Αυστρία, εάν θέλετε εξυγχρονισμό, θέλετε μια ανανέωση της οικονομίας, εάν θέλετε να έχετε κράτος δικαίου, δεν μπορείτε να το ανταλλάξετε για ένα πένι ή για ποσοστά. Πρόκειται για τα θεμέλια του πολιτισμού μας, όχι για το 0,1% πάνω ή κάτω. Αυτό οι Βρετανοί φίλοι μας θα το περιφρονούσαν. Ο κύριος... Ε, οι συντηρητικοί έχουν την άποψη ότι η χρηματοδότηση της ε, συνοχής ε, το 21 έως 27 θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο όπως από το 14 στο 20. Θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τη συγχρηματοδότηση και το υφιστάμενο επίπεδο πληρωμών. Εάν ε, περιστήλουμε την συνοχή είναι απαράδεκτο και αυτό θα μεταφερθεί σε προβλήματα μεταξύ δύο περιόδων προγραμματισμού. Επίσης έχουμε και το Brexit μπορούμε να ακυρώσουμε τις εκπτώσεις από το rebate από το 2021. Ε, όλες οι χώρες εισφορές θα πρέπει να, όλες οι χώρες θα πρέπει να πληρώνουν εισφορές βάσει των ίδιων κανόνων. Οι λόγοι για τις ε, εκπτώσεις δεν υφίστανται πλέον. Καμία χώρα μέλος δεν θα πρέπει να έχει υπερβολικό άχθος υπάρχουν χώρες αυτή τη στιγμή που πληρώνουν 5% ενώ άλλες χώρες ε, πληρώνουν πολύ περισσότερα. Ε, υπάρχει λοιπόν ένα ταμείο ε, μετασχηματισμού, αλλά δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται σε βάρος άλλων πολιτικών. Κυρία Μπιόρκ, ευχαριστώ πολύ. Πολύ προλαλήσαντες ζήτησαν περισσότερα κονδυλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ε, πρέπει να δούμε ε, ό,τι είναι το καλύτερο, καλύτερο για τον προϋπολογισμό με όρους ρεαλιστικούς. Δεν μπορούμε να ζητάμε απλώς περισσότερα κονδύλια Προφανώς, δεν, προφανώς θέλουμε ε, να καταπλημίσουμε την κλιματική αλλαγή, ε, χωρίς όμως να παραμελήσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές. Ε, σίγουρα δεν πρέπει να επενδύουμε πια σε τεχνολογίες μη φιλικές προς το κλίμα. Η ΚΑΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ε, μη χρηματοδοτηθούν άλλες πολιτικές. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να εξοικονομήσουμε από στρατιωτικές δαπάνες. Δεν θέλουμε επίσης κράτη-μέλη που δεν σέβονται τις βασικές αξίες και αρχές της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Κομίνη Ολιβέρης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για ένα καλύτερο προπολογισμό και μια πιο ισχυρή Ευρώπη και μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα. Χωρίς αυτά δεν θα καταρτήσουμε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό σύμφωνα με τις φιλοδοξίες μας. Θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια άμεση νομιμότητα. Ε, πώς θα φτιάξουμε ε, ένα δημοσιονομικό πλαίσιο που να είναι τόσο χαμηλό σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, για τις δημοσιονομικές προοπτικές 21-27 θα πρέπει να δώσουμε την προτεραιότητα στην ε, έρευνα, στην ενέργεια καθώς και τα ζητήματα δημοκρατίας, κοινωνικής ισότητας κλπ. Πότε θα έχουμε το θάρρος, το κουράγιο να οικοδομήσουμε ένα πραγματικό σύστημα ιδίων πόρων. Ο φόρος του άνθρακα θα πρέπει να εξυπηρετεί ένα νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γιατί από εκεί εξαρτάται το μέλλον της Ευρώπης. Η κυρία Χολμάιρ, 1,5 λεπτό. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητέ εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Ο τρόπος αντιμετώπισης του Συμβουλίου είναι άκρος προβληματικός. Λίγο συνοχή, λίγο κάπ, καμία φιλοδοξία για την επιστήμη, την έρευνα, λιγότερο Εράσμους, 1,0 είναι το μάξιμουμ, όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα, αλλά υποχρηματοδοτούμενα. Ο καθένας ε, ε, για τον εαυτό του και εγώ για τον εαυτό μου. Ε, αυτή είναι η προσέγγιση. Εμείς όμως ε, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την ε, ανάπτυξη ε, στις επιστήμες. Οι χώρες τη συνοχή πρέπει επίσης να βοηθηθούν να αναπτύξουν και να επενδύσουν στην έρευνα και τις επιστήμες. Αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν θα είμαστε πια ανταγωνιστικοί απέναντι στην Κίνα, ούτε απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν θα ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Πρέπει να έχω, θέτουμε καθήκοντα και να ανταποκρινόμαστε σε αυτά και να προβλέπουμε και τα απαραίτητα κονδύλια για να τα κάνουμε όλα. Αν θέλουμε να πληρώνουμε λιγότερα, να μας πει το Συμβούλιο τι θέλει να διαγράψει από αρμοδιότητες, από δραστηριότητες, ποιους οργανισμούς δεν θέλει, ε, τι δραστηριότητες θέλει να περιορίσει, αλλά να προβλέπει αύξηση δραστηριοτήτων και μείωση των δαπανών. Αυτό δεν γίνεται. Κλιματική αλλαγή πώς θα αντιμετωπιστεί χωρίς έρευνα και ε, ε ανάπτυξη ε, και, επιστήμες. Πρέπει επίσης να φύγουμε από την εθνική ε, θεώρηση των πραγμάτων και να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι στην προσέγγιση των προβλημάτων. Κύριε Σαντριό, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν έχουμε λιγότερο προπολογισμό με περισσότερες προσδοκίες, Έχουμε όλο και περισσότερε απογοητεύσει και λιγότερη Ευρώπη. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ενώ θα θέλαμε περισσότερη Ευρώπη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο συνεκτικοί και να έχουμε καλύτερη καθημερινότητα ω Ευρωπαίοι πολίτε. Αλλά για να έχουμε περισσότερη Ευρώπη πρέπει να επενδύσουμε στην Ευρώπη. Το διαπιστώνουμε όμω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο μηχανισμό για μια δίκαιη μετάβαση. Περιμένουμε τόσα πολλά από εκεί. Δεν, θέλει, δεν χρειάζεται να το σαμποτάρουμε από την αρχή. Υπάρχει η πολιτική συνοχή και η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική που πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τη στιγμή που υπάρχει ε, αύξηση τη θερμοκρασία του, του πλανήτη. Αυτό υπάρχει. Και το Green Deal πρέπει να είναι η χρυσή ευκαιρία για να αλλάξουμε βαθιά το οικονομικό μα μοντέλο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αποφασιστικό η ατζέντα των ε, ιδίων πόρων να συνδυαστεί με το Green Deal. Θα πρέπει η Ευρώπη να έχει τα μέσα για να μεταρρυθμιστεί. Με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή τη μάχη ε, θα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το Συμβούλιο δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών. Πέφτει σε, στα συμφέροντα του ενός και του άλλου. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με εγωισμούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακοσμητικές παρεμβάσεις ή μικρά μέτρα γελία ε, που ρυθμίζουν τα μικρά συνδυσιακά μας προβλήματα. Πρέπει να έχουμε ε, τα μέσα στο ύψος των πραγματικών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών. Αυτά τα μέσα τι σημαίνουν καταρχάς. Ένα πουδουπού, ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα προπολογισμό στο ύψο αυτών των προσδοκιών. Αλλά πρέπει να σας πω, σε εσά που συμμετέχετε στο Συμβούλιο, μην παίζετε μικροπολιτικά παιχνίδια, μην παίζετε μικρά παιχνίδια. Υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Για να μην πω είναι εντελώ ανεύθυνο πια. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, ο κύριος Νότεκ. Θα ήθελα να πω σε σχέση με τις ε, προτάσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνονται στι ε, προσδοκίες των πολιτών. 17% ε, των Ευρωπαίων πολιτών επιθυμούν επενδύσεις. Ε, τις ίδιες επενδύσεις όπως μέχρι τώρα στην, ε, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στην ε, πολιτική γεωργίας. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε αυτούς τους τομείς και είναι απαράδεκτο να μειωθούν οι επενδύσεις ε, στον τομέα της συνοχής, στη γεωργία και τις μεταφορές και ταυτόχρονα να αυξηθούν ε, οι χρηματοδοτήσεις άλλων τομέων. Θα πρέπει να είναι από τις χώρες μέλη που θέλουν να επενδύσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ακούει ε, τα αιτήματα των χωρών και να αφήσει τις χώρες να καθορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες. Βεβαίως είναι σημαντικό σημαντικό να γίνουν επενδύσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις βασικές υποδομές. Ο κύριος Κρούς για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, με εκπλήσει το ύφος, ο τόνος της συζήτησης, γιατί το θέμα λέγεται προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, του 2020 για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά τι κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς ε, ε κατηγορούμε το Συμβούλιο λέγοντας ότι δεν παρίσταται εδώ ο Σαλ Μισελ. Ε, ε, αυτό είναι επιζήμιο για τις ε, συζητήσεις. Θα πρέπει να επανέλθουμε ε, στο εξή. Τι θέλουμε ακριβώς. Το ζητούμενο εδώ είναι ξεκάθαρα το εξή. Έχουμε περιορισμένα κονδύλια και τα οποία, τα οποία θα πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε. Ας πάψουμε να δηλώνουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει ε, αν 1,7% είναι αρκετά χρήματα. Ένα λεπτό η κυρία Δεσούτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα επόμενα 7 χρόνια θα είναι κρίσιμα και θα καθορίσουν το πώς θα ζήσουν τα παιδιά μας σε αυτόν τον πλανήτη. Οι κοινωνίες μας θα πρέπει να κάνουν ένα ψηφιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό ε, σε έναν ε, οικολογικά αποδεκτό κόσμο. Ε, και κύριοι, ε, εδώ το ζήτημα αυτό είναι ο καθρέφτης του μέλλοντό μας. Ε, χρειαζόμαστε μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς ε, κατά ανάγκη αύξηση των ε, ιδίων πόρων. Μπορούμε να πάρουμε ιδίου πόρους από φορολόγηση μεγάλων οικονομικών συναλλαγών, κυροζήνης και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Γιατί εάν δεν συνειδητοποιήσουμε τις φιλοδοξίες του Green Deal, τότε οι πολίτες θα διαπιστώσουν ότι δεν γίνονται έργα υποδομών στις περιφέρειές τους ή ε, ε, χάνουν τις θέσεις απασχόλησης. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να αγκαλιάσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα και αυτό θα πρέπει κατά ανάγκη να αντανακλάται στον προϋπολογισμό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό θέμα. Οι Βρετανοί φεύγουν και πρέπει να δούμε την αναδιαμόρφωση των, του προϋπολογισμού. Ε, οι Βρετανοί υπήρξαν καθαροί χρηματοδότες και τώρα πρέπει να αυξηθούν ε, κατά, ε, στα 30, ε, ε, να, κατά 62% να αυξηθεί ο υπολογισμός. αυτά τα κονδύλια πώς θα βρεθούν. Δεν έχω δει κάποιον Πέρμαχο αυτών των ε, ε, προτάσεων. Α, βλέπω ε, ορισμένους να κάθονται χωρίς όμως να παρεμβαίνουν. Εγώ νοιάζομαι για τους Ολλανδούς πολίτες. Δείξτε θάρρος, ε, βάλτε βέτο όπως η Αυστριακή, πείτε ένα όχι ηχηρό για να επηρεάσετε έτσι τον προϋπολογισμό. Κύριος Φερέιρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, θα ε, πρέπει ε, να δούμε καθαρούς χρηματοδότες και μη. Ο χρόνος περνάει και πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι τα προβλήματα τους υπερβαίνουν. Καθυστερούν λοιπόν και αν υπάρχει καθυστέρηση χάνουμε ευκαιρίες. Τώρα αρχίζει ένας νέος γύρος. Θα πρέπει ο προϋπολογισμός να φροντίσει για τη μείωση των ανισορροπιών και των διαφορών. Η πολιτική συνοχή ε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν επαρκεί έτσι όπως είναι διαμορφωμένη για να ε, αντιμετωπίσει τις ανισότητες. Ε, αναφέρεται ότι η ε, νέες ε, πλούσιες χώρες, ε, ε, οι πλούσιες χώρες διαφωνούν σε σχέση με τα κονδύλια. Τώρα όμως θα πρέπει να φροντίσουμε για την Ευρώπη γενικότερα. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Σύντσις, ένα λεπτό. Κυρία Φόντερ Λάιν, μιλήσατε για τη χρηματοδότηση των διαφόρων πολιτικών. Η... Δεν μας είπατε όμως πώς χρηματοδοτείται στην Κροατία το σύστημα διάθεσης των αποβλήτων. Στην Κροατία χρειάστηκε να αναπτύξουμε 11 κέντρα διάθεση αποβλήτων, αλλά αυτό οδήγησε σε αύξηση του κόστους και της ρήπανσης. Γιατί αυτές οι αποτυχίες. Καταρχάς έχουμε τις κοινέ πολιτικές. Ας συγκρίνουμε τη Γερμανία και την Κροατία έχουμε τεράστιες διαφορές στο εισόδημα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτά που πληρώνει η Γερμανία. Δεν έχουμε επίσης ε, τα ίδια χαρακτηριστικά. Υπάρχει διαφθορά, όλα γίνονται λάθος στην Κροατία, δεν ανακυκλώνουμε τίποτα, όλα είναι δυσανάλογα, όλα είναι προς όφελος του κροατικού κατεστημένου για να βγάζει λεφτά. Και τελικά την ύφη την πληρώνει ο πολίτη, ο, ο Κροάτης πολίτης. Έτσι ζει ο πληθυσμό λόγω των υψηλών τιμών, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Λεβαντόσκι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Η ιστορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται. Αλλά στην περίπτωση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι κακό για το Κοινοβούλιο. Όταν ετοιμάστηκε το προσχέδιο προπολογισμού από την Κομισιόν το 2018, έκτοτε το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε μία άβολη κατάσταση. Δεν διαπραγματευόμαστε τα τομεακά project, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις αρχές αν δεν ξέρουμε τα νούμερα. Ε, και ο προπολογισμός αφορά τα νούμερα, δεν αφορά τις δηλώσεις. Πρόκειται περί αριθμών. Ο κύριος Σαλμισελ δεν είναι παρόν εδώ. Επομένως, δεν ξέρουμε αν οι ε, συναντήσεις του με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ε, κατηδίαν σε εξομολογητήρια οδήγησαν σε συμβασμούς ή όχι. Εάν ναι, τότε υπάρχει περίπτωση ε, να πετύχουμε και να πετύχει και η έκτακτη σύνδοση κορυφή τη 20 Φεβρουαρίου. Αλλά ποτέ δεν έχουμε πετύχει συμφωνία τον πρώτο γύρο. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση. Στην περίπτωση του 2014-2020 ε, όλα συμφωνήθηκαν στις 8 Φεβρουαρίου τότε μεταξύ των κυβερνήσεων και πέρασε η συμφωνία τελικά τον Ιούνιο. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν είναι ρεαλιστικά. Αν ε, τσακώνονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αυτό είναι πρόβλημα για την εικόνα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Λαρουτίχου για ένα λεπτό. Το 2012 ο Μάριο Ντράκη λέει ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι έτοιμες να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν την Ευρωζώνη. Και η κεντρική τράπεζα θα βάλει 2.600 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για τέσσερα χρόνια για να διασώσει την Ευρωζώνη και για και για να σώσουμε το κλίμα τι ποσά θα δώσουμε. Το να σώσουμε το ενιαίο νόμισμα ήταν πολύ σημαντικό προφανώς, αλλά το να διασώσουμε τον ενιαίο μας πλανήτη, την ενιαία μας ανθρωπότητα, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να πετύχουμε το Green Deal. Η ίδια η Επιτροπή λέει ότι λείπουν μεταξύ 300 και 500 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να σώσουμε το πλανήτη. Η λύση είναι να αναπτυχθούν ήδη πόροι προκειμένου να έχουμε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για το κλίμα. Όταν ήμουν μικρός ε, η φορολόγηση στα κέρδη ήταν 45%, σήμερα είναι 20%. Ε, ένα πραγματικό Green ε, Deal χρειάζεται μια αλλαγή εδώ και αυτό θα κριθεί τους επόμενους μήνες ο κύριος ε, Ντεσέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί που ξέρουν ότι δεν είμαι μόνο Γάλλος αλλά και γεωργός και πρώην εκπρόσωπος των γεωργών ε, θα, καταλα... θα καταλάβουν ότι, ε, ότι επιμένω στο βασικό διακύβημα που είναι η κοινή γεωργική πολιτική. είναι προς όφελος όλης της Ευρώπης. για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ε, χρειάζεται να γίνουν κάποιες θυσίες, ωστόσο θα ήταν σφάλμα και αυτό για τρεις λόγους όλες οι μεγάλες γεωργικές ε, δυνάμεις υποστηρίζουν τη γεωργία και εμείς θα πρέπει να βεσταθούμε σε αυτό το ύψος, όπως και οι άλλοι. Η οικολογική μετάβαση που βρίσκεται καθοδόν και το Green Deal δεν μπορούν να πετύχουν χωρίς μια κάπα που να έχει επαρκή κονδύλια. Ο προπολογισμό της κοινή αγροτικής πολιτικής εξαρτάται από την, ε, οδηγεί στην ποιότητα και στην ποικιλία της διατροφή μας και επίσης ε, οδηγεί στην την υποστήριξη των γεωργών. Ο προπολογισμό για τη γεωργία δεν θα πρέπει να μειωθεί. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ευχαριστώ που με καταλάβατε επίσης. Μπλε κάρτα ζητάτε κυρία Κουπίνη, αλλά έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την μπλε κάρτα. Ο κύριος Ντάβιτ ένα λεπτό. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ικανοποιείται με τη χαμηλή ανάπτυξη 1,1% στην Ευρώπη. Θα περίμενα λοιπόν σειρά μέτρων, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάει πίσω από την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. 40% του προϋπολογισμού θα έπρεπε να αφιερώνεται στην Πράσινη Συμφωνία για να μην καταστραφεί η οικονομία μας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημαίνουν ε, α, όμως ε, ότι θα υπάρξει επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα γιατί οι παλιές τεχνολογίες θα εγκαταλειφθούν, πράγμα που θα οδηγήσει σε στασιμότητα και υπάρχουν πολλές ομάδες πίεσης όπως μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που παίζουν ρόλο. Βλέπετε λοιπόν ε, πώς, πώς ε, εξελίσσονται τα πράγματα. Δηλαδή ε, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την μετανάστευση αντί να βοηθήσουμε τις αγροτικές μας περιοχές και την Ήπεθρο. Είπατε ότι θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις, ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις, αλλά ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ. Ο κύριος Κούσμιουκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Ροπέ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία. Η απόφαση για το πολιετές δεν αφορά χρήματα, αλλά στόχους. Δεν ε, φροντίζομαι για τις συνθήκες διαβίωσης. Ε, η συνοχή έχει περικοπεί σημαντικά θα την ανεχθούμε αυτή την κατάσταση ε, όταν κάποιοι αγρότες αντιμετωπίζονται ως ε, ε, κατώτεροι. Νομίζω ότι είναι σαφές το όχι. Ποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί για μας, εκείνοι των κρατών μελών ή οι κοινοί μας στόχοι. Αυτή η ερώτηση αφορά τη συζήτηση για το εύρος τη συνεισφορά των κρατών μελών στον προπολογισμό. Βεβαίω έχουμε νέε προκλήσει, αλλά χρειάζονται και νέα κονδύλια για τη χρηματοδότησή του. Δεν αφαιρούμε μόνο χρηματοδότηση από συγκεκριμένους τομείς, αλλά έχουμε και μια κοινή συμφωνία ε, που λέει ότι δεν πρέπει να τη συνεχίσουμε πια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, Επίτροπε, οι περικοπές 10% ε, στην ε, πολιτική συνοχή και στην ΚΑΠ απορρίφθηκαν από τη ε, θέση που υιοθετήθηκε στην Πορτογαλία από τις χώρες συνοχής. Απορρίφθηκε από αυτές τις χώρες. Ίσως θα πρέπει να μειώσουμε τα rebates, τις εκτόσεις και να βρούμε νέους ίδιους πόρους. Ένας συμβασμός στο Συμβούλιο είναι δυνατός, υπό τον όρο όμως ότι δεν διαπραγματευόμαστε πια μέσα, μέσω της οπτικής των ε, πληρωτών και εκείνων που εισπράττουν. Λαμβάνοντας υπόψη όμως τα ωφέλη των διαφόρων χωρών από τις ε, κεφαλιακές ροές και από την ενιαία αγορά. Οι καθαροί πληρωτές εποφελούνται από τη συμμετοχή ε, στην ενιαία αγορά. Γερμανοί κερδίζουν 200 δισεκατομμύρια, ενώ πληρώνουν το 27% στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και άλλες δυτικές χώρες ε, εποφελούνται από τη συμμετοχή στην ενιαία αγορά. Έχουν ε, μέσω των κεφαλαίων και των κερδών τους. Μόνο ε, έτσι, αν τα δούμε όλα συνολικά, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμβασμός. Ο κύριος Ρέσλερ. συνάδελφοι, ε, μια πετυχημένη Ευρώπη στις νέες γενιές είναι δυνατή μόνο με ισχυρές επενδύσεις στις επιχειρήσεις, στην έρευνα, στην νεολαία, στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να προβούμε σε μια ποιοτική προσαρμογή της υπήρου, της υπήρου μας ε, σε σχέση με τη ψηφιακή επανάσταση. Αλλά επίσης θα πρέπει να εξοπλιστούμε ε, όσον αφορά την κούρσα για τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με ισχυρότερους αντιπάλους. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να εξισορροπήσει, να μειώσει τις ε, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών. Γιατί αυτό, ε, αυτός είναι ένας βασικός στόχος ε, των συνθήκων. Εκεί επισημαίνεται ρητά ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες οι οποίες ε, πάσχουν από δημογραφικές ε, δυσκολίες και θα πρέπει να κάνουν μια βιομηχανική ε, αλλαγή, μετάβαση έχει έρθει πλήρωμα του χρόνο προκειμένου ο ευρωπαϊκό προπολογισμό ακριβώ λόγω τη συνοχή αλλά και ακριβώ λόγω τη ίση όλων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα ευρωπαϊκά εργαλεία υποστηρίζουν αυτές τις περιφέρειες. Λοιπόν, αφέ, ένα λεπτό. Την επόμενη εβδομάδα το Ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει ένα αποφασιστικό θέμα. Τι πόρους θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 μέχρι το 2027 για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας και να δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες μια κοινωνία πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά, πιο δίκαιη, πιο ασφαλή, πιο μοντέρνα. Το Κοινοβούλιο ζήτησε ένα φιλόδοξο προπολογισμό. Μέχρι στιγμή η απάντηση των κυβερνήσεων ήταν ανεπαρκή. Από τη μία δίνουμε νέα καθήκοντα στην Ευρώπη, με καθήκοντα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσει μόνε. Από την άλλη όμω δεν βάζουν οι κυβερνήσει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή θέλουν να κάνουν περισσότερα, θέλουν η Ευρώπη να κάνει περισσότερα αλλά με λιγότερου πόρου χρησιμοποιούν ουσιαστικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ω τον καλύτερο αποδιοπομπαίο τράγο για ό,τι πάει στραβά. Εδώ δεν δικαιολογείται, συνάδελφοι, ένα προπολογισμό, αλλά η ίδια η αξιοπιστία τη Ένωση. Ζητάμε από την Προεδρία του Συμβουλίου να στείλει το μήνυμα του Κοινοβουλίου στους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων. Θέλουμε μια αντιστροφή, των τάσεων. Ε, θέλουμε να ανοίξει ο διάλογος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόρβαλτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ίσως θα έπρεπε να ρωτήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Πρόκειται για την πρόκληση ε, της δημιουργίας ενός νέου οικολογικού βιομηχανικού συστήματος. Δεν είναι επιστημονική φαντασία αυτό, είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πρωτίστως έναν ε, προϋπολογισμό συμβατό με το Παρίσι, έναν προϋπολογισμό με βάση την Πράσινη Συμφωνία για τα επόμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό για την έρευνα που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές προκλήσεις. Και αυτός ο προϋπολογισμός για την έρευνα θα πρέπει να είναι συμβατός και με τους προϋπολογισμούς για την έρευνα των κρατών μελών. Πρόκειται για περισσότερη και όχι για λιγότερη Ευρώπη. Κύριε Μπιτζότο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύετε ότι οι Ιταλοί είναι ηλίθιοι. Πιστεύετε ότι μπορείτε να τους κοροϊδεύετε επάπειρον. Ως πότε θα πρέπει να υφίστανται τις αποφάσεις της Ευρώπης. Νομίζω ότι αγαπητοί γραφειοκράτες ε, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Είναι ε, κουρασμένοι που τους κλέβετε κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, όλοι έχουμε κουραστεί να βλέπουμε πώς η Ευρώπη κλέβει τα λεφτά μας και τα δίνει στην Τουρκία του Ερντοάν για να επαναπατρίσει με λαθρομετανάστες στα σπίτια τους. Αυτό είναι ντροπή. Αλλά προετοιμάζεται ακόμα χειρότερα. Τα επόμενα αυτά χρόνια θέλετε ναι, να επιβάλλετε νέο φόρο, τον πληρώνουν οι πολίτες μας, που τον κρύβεται με ονόματα όπως οι διπόροι. Και επίσης θέλετε να μας ε, εξαπατήσετε, να μας κλέψετε. Προσοχή, προσοχή. Τέλειωσε η υπομονή των Ιταλών. Θα κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε τις τρέλες αυτής της Ευρώπης. Η κυρία Βρυσιόνοβα, ένα λεπτό. Καλημέρα σας, ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι από την Τσεχία, μια χώρα που είναι φίλη της συνοχής, όπως λέγεται. Εγώ όμως προτιμώ την αρχική πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όχι την πρόταση του Κοινοβουλίου. Γιατί οι μεγαλύτερες δαπάνες που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνουν περισσότερες συνεισφορές. Οι καθαροί συνεισφέροντες δεν θέλουν να αυξήσουν την εισφορά τους και ένας από τους μεγαλύτερους ε, συνεισφέροντες εγκατέλειψε την Ένωση την περασμένη εβδομάδα οι ίδιοι πόροι θα επαρκούν. Ακούσαμε πολλά για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι οι ίδιοι πόροι δεν είναι καλός τρόπος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπερκράτος. Ε, είναι ε, ένα οργανισμό που αποτελείται από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται την βούληση των κρατών μελών και δεν μπορεί να φορολογούνται άμεσα οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ε, ε, ε, στηρίξουμε περισσότερο τις υποδομές και την καινοτομία. Το, η τελευταία εκδοχή του προϋπολογισμού νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσει πίσω προς τις εκδοχές της ε, Κομισιόν. ένα 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, ε, βλέπουμε πολλούς νέους που ενδιαφέρονται για το έρασμο, την έρευνα, την ανάπτυξη, υπάρχουν οι στρατιώτες μας που θα πρέπει να τους δώσουμε απαντήσεις σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, την πολιτική άμυνας. Ο Σάρλ Μισελ λέει ότι στις 20 Φεβρουαρίου θα αφήσει τους ηγέτες να φύγουν μόνο αν βρεθεί λύση. Πρέπει να λάβει και εμάς υπόψη. Τα κράτη συνοχής, αυτά που ωφελούνται δηλαδή περισσότερο από την πολιτική συνοχής, θέλουν περισσότερη ευελιξία για την εφαρμογή του συστήματος. Αυτό είναι καλό, αλλά οι πόροι δεν επαρκούν. Αν χρειάζεται περισσότερη ευελιξία, αυτό είναι καλό, αλλά δεν υποκαθιστά τα κονδύλια που λείπουν. Ε, δεν θα ε, παίξουμε παιχνίδια εδώ ότι ε, θα ε, σας, ε, θα δεχτούμε λιγότερα ε, κονδύλια αλλά θα δεχ, μας δώσετε περισσότερη ευελιξία. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κοινή προσέγγιση. Ε, ελπίζω στις 20 Φεβρουαρίου να βρεθεί λύση μετά από την πρόσκληση του Σαρλ Μισελ. Τώρα το θέμα του, του, του, του των κονδυλίων που θα προβλέψουμε για τον προϋπολογισμό αυτό είναι στο επίκεντρο. Ευχαριστώ. Πλάμ, ένα λεπτό. Κυρία ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ένα στέρεο προπολογισμό, ο οποίο λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες που έχουμε να επιτρέψουμε την ανάπτυξη που είναι τόσο αναγκαία ε, στο επίπεδο των χωρών μελών, αλλά θα πρέπει να είναι και μια απάντηση στις νέες προκλήσεις. Πιστεύω ότι ο προπολογισμό δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια μαθηματική άσκηση, αλλά θα πρέπει να είμαστε συνεπεί προ το ευρωπαϊκό εγχείρημα, για παράδειγμα πολιτική συνοχή. Το Κοινοβούλιο ήδη απεφάνθη εδώ το, δεν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το Ταμείο Συνοχής με νέες ε, πρωτοβουλίες όπως είναι το Ταμείο Μετάβασης που βεβαίως θα πρέπει να έχει όλους τους αναγκαίους πόρους προκειμένου η μετάβαση αυτή να είναι δίκαιη. Εάν δεν αναφερθούμε στις ε, μεταφορές, ο Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης ε, εδώ αποφάνθηκε και το Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να μειωθεί επίσης η χρηματοδότηση, γιατί ε, εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία μας όσον αφορά τις νέες προκλήσεις και τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρακαλώ συνάδελφοι να είστε πιο ευέλικτοι, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν το λόγο στο πλαίσιο του Catch the Eye. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γαρινακάνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη ε, αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή κρίση. Ε, τα λαϊκιστικά κόμματα πολλαπλασιάζονται. Ε, η όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη υπάρχει μια στασιμότητα ε, τι γίνεται με την Τραπεζική Ένωση. Με, την, τον Brexit χάνουμε ένα βασικό μέλος. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια υπαρξιακή κρίση και έναν προπολογισμό ο οποίος είναι ο πιο χαμηλός ε, στην ιστορία μας. Έχουμε πολλές προκλήσεις και δεν έχουμε τα, τους αναγκαίους πόρους να, να τις αντιμετωπίσουμε. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται για τους καθαρούς συνεισφέροντες, ε, για αυτούς που παίρνουν πόρους. Αλλά η συζήτηση αυτή δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ιδίων πόρων, το οποίο να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής και φοροδιαφυγής. Το κοινοβούλιο αυτό δεν θα εγκρίνει μία συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μονσερά, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα ε, δεν θα είναι πιο ισχυρό με μια αποδυναμωμένη Ευρώπη. Τα νέα που μας φάνουν από την Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι καλά. Ε, μείωση της ΚΑΠ, ε, μείωση του Κοινωνικού Ταμείου κλπ. Δηλαδή αποκρινόμαστε, αποκρίνουμε από την Ένωση εκείνους που πιο πολύ την έχουν ανάγκη. Οι Ισπανοί επίσης πάσχουν ε, γιατί από τη μία πλευρά τους ζητούν αύξηση ανταγωνιστικότητας, από την άλλη δεν υπάρχει αναγκαία χρηματοδότηση της αγροτικής πολιτικής. Ή η νεολαία στην Ισπανία ε, η οποία έχει τρομερά υψηλά ποσοστά, 30% από τη μία υπάρχουν αυτές οι ανάγκες, από την άλλη μειώνονται οι πόροι. Ή ε, η ψηφιακή πρόκληση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κατάσταση πέθρου. Ε, δεν είναι συνεπές να λέμε ότι βοηθάμε τις περιφέρειες με λιγότερους πόρους για τη συνοχή. Ε, θα πρέπει τα μέλη να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ε, το Λαϊκό Κόμμα στην ε, Ισπανία δίνει μάχες που χάνονται και οι σοσιαλιστικές ε, κυβερνήσεις τελικά γυρνούν στην Ισπανία με άδεια χέρια. Τα διαφορετικά ταμεία, η μειώση των διαφορετικών ταμείων για τα ταμείων συνοχής θα πλήξουν καθοριστικά την Ισπανία. Θα πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη για την ενίσχυση των περιφερειών και της υπαίθρου. Ένα λεπτό, κύριος Μπέρκβιστε. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς. Έχουμε τόσο μεγάλη ευκαιρία εδώ. Μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις για μια ειρηνική ε, ανάπτυξη και ευημερία. Ε, όλα δείχνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία για να βελτιωθούν τα πράγματα γενικότερα. Σίγουρα υπάρχουν ε, κίνδυνοι, υπάρχουν ε, ο κίνδυνος του λαϊκισμού, του εθνικισμού, υπάρχουν ενδιασμοί. Αν υποκύψουμε θα χάσουμε αλλά κατά τα άλλα είμαστε η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μια τεράστια περιφέρεια με ε, τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν να αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις και για το κλίμα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στους εθνικισμούς. Ο Φρανσουά Μιτεράν είχε πει ότι ο εθνικισμός σημαίνει πόλεμο. Ε, μπορεί να ισχύει αυτό, να είναι πόλεμος ε, και για το μέλλον. Ε, πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες της ειρήνης και της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Η κυρία Νάκτεγκάλ, ένα λεπτό. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα περνάει από μια φάση make or break. Πρέπει να αναρωτηθούμε θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του χτες ή πρέπει να, ε, έχουμε, ε, να προσπίσουμε τα κοινά συμφέροντα όλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να να προσπισουμε τα κοινα συμφεροντα ολων η ευρωπαικη ενωση θα πρεπει να αντιμετωπισει τις κοινέ προκλήσεις. Μετανάστευση, ασφάλεια, κλίμα. Αυτά ζητούν οι πολίτες από την Ένωση. Και γι' αυτό χρειάζεται λογοδοσία προβλέψιμες ε, πολιτικές ε, δεν μπορούμε να ε, λειτουργούμε όσο αν έχει μικρύνει η Ένωση. Οι χώρες θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφο επίπεδο ανάπτυξης και να μπορούν και να αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχει διαφθορά σε μια χώρα ή αν ε, καταστρατηγείται το κράτος δικαίου, ε, τότε θα μπορεί να μην χορηγούνται κονδύλια, να υπάρχει μια σύνδεση. Ε, δεν θα πρέπει να χωριστούμε, να διαιρεθούμε σε Ευρώπη του Βορρά, του Νότου κλπ. Αλλά να προχωρήσουμε ενωμένοι. Ο κύριος ε, Ντόιτς, μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, η φιλανδική κυβέρνηση ε, τα, τα μπέρδεψε τα πράγματα. Η Φιλανδική Προεδρία, και εδώ ε, επιλέγω ήπιο χαρακτηρισμό, ε, ανταποκρίθηκε με υποβέλτιστο τρόπο και τώρα απέχουμε πολύ από μια συμφωνία πολύ πιο μακριά από μια συμφωνία από ότι είμαστε επί Αυστριακής ή Βουλγαρικής Προεδρίας. Η Κροατική Προεδρία τώρα έχει ένα τεράστιο καθήκον. Η Φιλανδική Προεδρία παρουσίασε ένα άδικο σύστημα, το οποίο ε, έχει λογική που δεν στέκει. Η λογική λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει και να βελτιωθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είναι άδικο